Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική T17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 179 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 181 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται R34, απευθείας πάμε στο R34, άρχεται η ψηφοφορία. R34. R34 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. R35. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περάμε στο R36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. R37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 197. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική R38 άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική R39 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 207 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία υπαριθμών 212. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Περνάμε στο 2.11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική R40, άρχεται. R40. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. R41, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται, τροπολογία 227, άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική R42, άρχεται. Πέρας, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 238, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απερίφθη. Συμβαστική R43, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική R44, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβετροπολογία 254. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην συμβαστική R45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική R47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 275. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απερίφθη και περνάμε στη συμβαστική R48. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. R49 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, 285 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική R50 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 298 άρχεται η ψηφοφορία. 288, συγγνώμη, πέρας ψηφοφορίας ε, ε, απορρίπτεται 300 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβαστική σε ΙΟΕ 31 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 309. Τροπολογία 309. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 310. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σε 32. Άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 320. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 321. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 322. Άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 324. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 323. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 325 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίες απορρίπτεται. 326 άρχεται ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική σε 33 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική σε 34 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 331 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 332, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 333 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 334 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 335 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 339 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 336 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 335 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 338 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 450. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 340. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 341. Απορρίπτεται. 342. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 343. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 344. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 441. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 345. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 347. Καταπίπτει, λέει πρόεδρος. Άρα πάμε στη σε ΣΕΙΟΕ 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 349, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 350 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμό 351. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 352. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική σε 36. Ε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 358. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 359. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 360. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σε 37 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία εγκρίνεται. 369 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 368. Το πρώτο τμήμα. 368. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα 368. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Η γραμματεία εξηγείται ότι όταν ε, είναι χωριστή ψηφοφορία θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Και εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται από συνήθεια. Δεν ξέρω, λέει ο πρόεδρος. Να συνεχίσουμε, λέω, ε, όσο το, το ε, ε, το κείμενο όταν δεν είναι χωριστή η ψηφοφορία, άρα εγκρίνεται. Όλοι, άρα είχαμε σφάλει. Εγκρίνεται, μου λέει η γραμματεία. Εντάξει, αυτό δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά... 370 και 371 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 372 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική σε 38 άρχεται η ψηφοφορία σου ψηφοφορία εγκρίνεται. 381 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Εγκρίνεται. 382 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 383. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σεβαστική ΣΕΙΟΕ 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 390 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΣΕΙΕ 40 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 396 ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτωτε. Τροπολογία 397. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίναμε την 397, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, ακούγεται από κάτω. Θέλετε να επαναλάβουμε, λέει η Επαναλαμβάνουμε την 397. Ξανά την 397 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 398. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική CIE 41. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 404. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 405. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 406. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Α, απορρίπτεται. 407. Άρχεται η ψηφοφορία. 407. Απορρίπτεται. 409. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 408. Ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 410. Ξεκινάμε. Πέρα τούτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. CIE 42. Ξεκινάμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΒ12. Ξεκινάμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 424. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 425. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 400. συμβιβαστικη ΕΒ13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΕΒ14. Ξεκινάμε. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 435, ξεκινάμε. Έλλειξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 436. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 437. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 438. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 439. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. 440. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 434. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 442-443 είναι ταυτόσιμες και ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνονται. 444. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 451. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική ΕΒ15, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΒ16, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΒ17. Ξεκινάμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 464. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική CTF 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική CTF 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 470. Άρχεται η ψηφοφορία.

Πέρας. Εγκρίνεται. 473. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική CTF 12. Ξεκινάμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική CTF 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 482. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 484. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται επί της 484. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 485. Πάμε στο CTF 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 490. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 491. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 492 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε 534. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική ED3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 540. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 541. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 542. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 543. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 543. Συμβαστική ED4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. d ED5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 554. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 555. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 556. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 557. Απορρίπτεται. 558. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 559. Ψηφίζουμε. Τέλος. απορρίπτεται. Πεντακόσια εξήντα. Ψηφίζουμε. Θα επαναλάβουμε αυτή την τροπολογία. Την 569 και την 560. Υπήρχε ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο. Μπορείτε να μετρήσετε παρακαλώ. Θα επαναλάβουμε. Ξαναρχίζουμε λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναψηφίζουμε την τροπολογία 559. Ξεκινάμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 560. Ξεκινάμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Ξεκινάμε. Τροπολογία 561 ψηφίζουμε, λέει ο Πρόεδρος. 561. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, 562. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 563. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 564 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 565 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική. V6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. V7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 577. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απερίφθη. Τροπολογία 579 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 580 άρχεται. Πέρας απερίφθη. Συμβιβαστική 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 582 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απερίφθη. 585 άρχεται. Πέρας, απερίφθη. 586 άρχεται πέρας απερίφθη 587 άρχεται πέρας εγκρίνεται 588 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 589 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 591 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη 592 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 593 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται 594 άρχεται πέρας απερίφθη μια και το προήμιο έχει ήδη γίνει δεκτό το επόμενο τμήμα καταπίπτει και πάμε απευθείας στη συμβιβαστική FR1 άρχεται Πέρας εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική FR2. Όχι. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής FR2. Ψηφίζουμε για το FR2 τρία, λέει η πρόεδρος. Να ψηφίσουμε το FR3 και μετά θα επαληθεύσουμε αν τα κάναμε σωστά, λέει η πρόεδρος. C'est ça vous le sent ou pas Parce que ça c'est l'indication après.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 Παρ' όλα αυτά πρέπει να ψηφίσουμε και τη συμβαστική FR2. Ξαναλέω λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε και την συμβαστική FR2. Il a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 Λοιπόν, έχουμε ήδη εγκρίνει την FR3 και περνάμε στην FR4. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής FR4. Το 3 το έχουμε ψηφίσει. Δεν ξαναψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 613. Άρχεται η ψηφοφορία. ε, απερίφθη. Τροπολογία 608, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 609, άρχεται 609 και 590 από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και απερίφθη. Τροπολογία 611. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 611. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία υπερθυμών 18, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απερίφθη. Τροπολογία υπαριθμό 616, άρχεται η ψηφοφορία. Επί της 616. Πέρας. Απερίφθη. Τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. Είστε έτοιμοι. Are you ready? Άρχεται η ψηφοφορία. Ας περιμένουμε λίγο. Voilà. Le vote est clos. 23 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και βεβαίως συγχαρητήρια στις δύο συνεισηγήτριες και ε, μπράβο και συγχαρητήρια και έβγε στους σκιώδεις και σε όλους. Δουλέψαμε πάρα πολύ γρήγορα, κερδίσαμε ένα, ε, μία ώρα και 15 λεπτά. Η Μόνικα θέλει να μιλήσει. ήθελα να πω, απλώς λέει η κυρία Χολμάιερ, ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ και εξ ονόματος της Helga Stevens ε, και της υποφαινομένης. Να σας ευχαριστήσω όλους γιατί δουλέψαμε σκληρά, δουλέψαμε πολύ. Ποτέ δεν είδα μέχρι τώρα μία τόσο καλά δομημένη και τόσο καλά συντονισμένη ψηφοφορία και τόσο καλό κατάλογο ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε τη Γραμματεία γι' αυτό και ευχαριστούμε βεβαίως και όλους τους συμβούλους μας και όλο το σύστημα για την τρομερή βοήθεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ λέει η Πρόεδρος και πριν τελειώσουμε θα ήθελα να σας ζητήσω να σημειώσετε στις ατζέντε σας ε, αυτό το ε, κέρασμα που θα οργανώσουμε στις Βρυξέλλες, το κέρασμα της φιλίας θα γίνει στις Βρυξέλλες ε, μετά από τόσο μεγάλη και πολλή δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν σημειώστε το. Παρακαλώ πολύ να είστε όλοι εκεί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστεί η Πρόεδρος Ευγενός τους Διερμηνείς και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί.